Αγαπητοί συνάδελφοι, η ελευθερία των μέσων ενημέρωση και ο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση είναι μια βασική αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Τουρκία είναι μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να υπάρχουν διαπραγματεύσει και πρόοδο πρέπει να υπάρχει αμοιβαία πρόοδο. Θέλουμε να λάβουμε το θέμα της Τουρκίας στα σοβαρά, οπότε είναι απαραίτητο να τονίσουμε πότε υπάρχουν πρόοδοι, αλλά όταν υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Αυτά τα γεγονότα σε σχέση με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία δεν είναι καινούρια. Εμείς με μεγάλη έκπληξη είδαμε τις ε, ε, συλλήψεις εναντίον δημοσιογράφων και εναντίον μέσων ενημέρωσης στο παρελθόν με την ευκαιρία των διαδηλώσεων στο Γκεζί Πάρκ και χθε είδαμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες ενέργειες και νιώθουμε βαθιά ανησυχία γιατί με τον τρόπο αυτό διακόπτεται ο πρόεδρος.